περιβαλλοντικές πτυχές, βιολογικές πτυχές, αλλά οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Πέρας λοιπόν της κοινή συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί στις 11.30. Οπότε συνεχίζουμε με την επόμενη κοινή έκθεση, μάλλον κοινή συζήτηση που αφορά την ε, τις πληροφορίες για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Ε, θέλω να καλωσορίσω τον Επίτροπο Ντάλη. Δίνω το λόγο για τέσσερα λεπτά στον εισηγητή, τον κύριο Φιέλνερ. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, επιτέλους έφτασε στην Ολομέλεια η νέα νομοθεσία που αφορά τις πληροφορίες για τα φάρμακα ενδεχομένως είναι το τελευταίο και το πιο αμφιλεγόμενο ε, κομμάτι του πακέτου των φαρμάκων. Πριν από ένα χρόνο ποτέ δεν θα πίστευα ότι θα φτάναμε από κοινού στην Ολομέλεια με τόσο μεγάλη ενότητα, συνένεση όπως τώρα. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι δούλεψαν εξαιρετικά υποδομητικά και έδειξαν διάθεση συμβιβασμού. Γι' αυτό καταφέραμε να συγκεντρώσουμε τόσο μεγάλη υποστήριξη για την έκθεση αυτή στην Ολομέλεια. Δεν είναι απλώς και μόνο η επιθυμία, η προθυμία για συμβιβασμό, αλλά πιστεύω ότι όλοι καταλάβαμε ότι όλοι εδώ στο Κοινοβούλιο θέλουν να προχωρήσουμε προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή να έχουμε καλύτερες και πιο ευκολότερα προσβάσιμες πληροφορίες ε, για τα φαρμακευτικά προϊόντα υπέρ των ασθενών πράγμα που να μην αποτελεί ούτε διαφήμιση ούτε κρυφή διαφήμιση υπέρ των φαρμάκων. Τρίτον, θέλουμε τις πληροφορίες που απευθύνονται στους ασθενείς και οι οποίες ε, παρέχονται από τις ε, εταιρείε να ελέγχονται σωστά και να επικυρώνονται από τις αρμόδιες αρχές. Όλοι ε, συμφώνησαν με αυτές τις αρχές και γι' αυτό ήταν εύκολη η συμφωνία. Θεωρήσαμε ότι ήταν σε κάποια σημεία αναγκαίο να αναδιατυπώσουμε τις προτάσεις της Κομισιόν Θέλω να αναφερθώ κυρίως σε πέντε σημεία. Πρώτον, αλλάξαμε την σκοπιά της νομοθεσίας. Δηλαδή, πλέον δεν αφορά το δικαίωμα των εταιριών να διανέμουν πληροφορίες. Όχι, αφορά το δικαίωμα των ασθενών να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Αυτό είναι το βασικότερο σημείο. Είναι καθήκον των εταιριών να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες. Δεύτερον, ε, εξετάσαμε τις διάφορες εξαιρέσεις για να διαπιστώσουμε ότι δεν θα, υπήρξαν, δεν θα υπήρχαν παραθυράκια για κρυφή διαφήμιση. Τρίτον, εξασφαλίσαμε ότι οι πληροφορίες που παρέχουν οι φαρμακευτικές εταιρείε επιτηρούνται σωστά και είναι αξιόπιστες. Διότι κάποια στιγμή στην διάρκεια αυτή τη αλυσίδα χρειάζεται κάποιο αποτελεσματικό έλεγχο. Τέταρτον, εξασφαλίσαμε όλε οι πληροφορίε που προέρχονται από τι φαρμακευτικέ εταιρείε είναι πληροφορίες που θα πρέπει να ζητούν οι ασθενείς. Ποτέ δεν θα πρέπει να λαμβάνει κανείς πληροφορίες από μια φαρμακευτική εταιρεία χωρίς να τη ζητά. Δεν το, ε, έχουμε το μοντέλο της πρόθεσης δηλαδή της διαφήμισης από τα μέσα ενημέρωσης. Και τέλος θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει οι εταιρείε να είναι το τελικό σημείο της αλυσίδας πληροφοριών. Σε πολλές χώρες οι πάροχοι ε, περίθαλψης πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να παίξουν τον ρόλο που τους αναλογεί. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι γιατροί προς τους ασθενείς αποτελεί συγκεκριμένη εξαίρεση από την όλη αυτή διαδικασία. Δηλαδή ένας ε, γιατρός στη Σουηδία δεν μπορεί να ε, παράχει, παράσχει πληροφορίες ε, ε, στα αγγλικά σε έναν ασθενή που δεν καταλαβαίνει σουηδικά παρά μόνο αν υπάρξουν κάποιες ε, εξαιρέσεις. Γιατί βεβαίως τα αγγλικά δεν είναι επίσημη γλώσσα της Σουηδίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, του Συμβουλίου Υπουργών. Δυστυχώ δεν παρίσταται το Συμβουλίο Υπουργών εδώ σήμερα, αλλά δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στα επιχειρήματά του. Μέχρι στιγμή όμω δεν ε, πήραμε πάρα πολλέ λεπτομέρειε από το Συμβούλιο θέλαμε περισσότερες. Παρά τα αυτά, εδώ στο Κοινοβούλιο εμείς καταφέραμε να επιτύχουμε μια συμφωνία, σχεδόν ομοφωνία. Και πιστεύουμε ότι με περαιτέρω δουλειά θα φέρουμε και το Συμβούλιο πιο κοντά στις απόψεις μας. Δεν θέλουμε όμως αυτό να οδηγήσει απλά και μόνο σε, εξοικονο... σε οικονομίες, σε εξοικονόμηση ε, δαπανών. Βεβαίω ε, θα ε, εξοικονομηθούν χρήματα, αλλά όχι σε βάρος της ενημέρωσης των ασθενών. Να εργαστούμε, να προσφέρουμε καλύτερη ενημέρωση στους ασθενείς της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Φέλνερ. Το λόγο έχει ο Επίτροπος Ντάλι. <coughs> Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Κατά τη διάρκεια της ακροάσεώς μου, ε, όταν ήμουν υποψήφιος επίτροπος, ξεκαθάρισα ότι η ενημέρωση των ασθενών αποτελεί για μένα ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Οι ασθενείς ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την υγεία τους και την ε, ευημερία τους. Όμως η πληροφορία για τα φάρμακα στην Ευρώπη είναι πολυπίκυλη και θα έλεγε κανείς και άδικη εάν οι ασθενείς, το αν οι ασθενείς θα πάρουν τις ε, αρμόδιες ε, πληροφορίες εξαρτάται από τη γλώσσα, από την δυνατότητα να χειριστούν ε, την πληροφορική και ίσως και από τη χώρα αυτό είναι μια ανισότητα που δεν μπορεί να παραμείνει. Η βασική φιλοδοξία της πρότασης της Κομισιόν εξακολουθεί να είναι ε, η ίδια και δικαιολογημένη. Και χαιρετίζω το Κοινοβούλιο και κυρίως τον εισηγητή, τον κύριο Φιέλνερ, που ανέλαβε να προωθήσει αυτή τη σημαντική πρόταση. Όμως πιστεύω, όπως επίσης υπογράμμισα κατά τη διάρκεια τη ακροάσεώ μου ότι το θέμα αυτό πρέπει να το δούμε από τη σκοπιά των ασθενών. Πρέπει να διαρωτηθούμε ποιες είναι οι πληροφορίες χρειάζονται οι ασθενείς και όχι ποιες θα πρέπει να προσφέρουν οι εταιρείε. και δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε ή να γλιστρήσουμε προς άμεση καταναλωτική διαφήμιση που δεν χρειάζονται οι ασθενείς. Βεβαίως και χαιρετίζω τις θέσεις του Κοινοβουλίου γιατί επιτρέπει στην Κομισιόν να αποδεχτεί πολλές από τις βασικές τροπολογίες σας όταν θα παρουσιάσουμε τις τροποποιημένες προτάσεις μας μεταξύ των οποίων την υποχρέωση δημοσίευσης των πληροφοριών το θέμα των ποιον, ποιες πληροφορίες καλύπτονται, το θέμα της ε, ε μετάδοσης των πληροφοριών μέσω μιας αλυσίδας και, της, ε, ε, και του ελέγχου των πληροφοριών. Βεβαίως είμαι υπέρ της ε, της ε, τροπολογίας ε, για το ότι πρέπει να παρέχονται πληροφορίες δεύτερον όσον αφορά το ποιο, ποιες πληροφορίες δεν θα πρέπει, συμφωνώ και εγώ, να υπάρχει συγκριτική ε, παράθεση πληροφοριών γιατί αυτό μπορεί να θεωρηθεί πρόθεση. Οι πληροφορίες πρέπει να αφορούν και τους ασθενείς και τους παρόχους υγείας αλλά λόγω της κατάχρησης που μπορεί να γίνει για λόγους διαφήμισης χρειάζεται στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη στον τομέα της αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας. Επίσης συμφωνώ ότι οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν τις πληροφορίες που προσφέρει ο κλάδος και όχι τρίτη όπως επιστήμονες ή δημοσιογράφοι. Γνωρίζουμε όμως υπάρχει μια, μια γκρίζα ζώνη που αφήνει περιθώριο κατάχρηστης. Γι' αυτό θα πρέπει αυτές οι πλευρές να κάνουν δήλωση για τυχόν οικονομική ενίσχυση από τη βιομηχανία. Όσον αφορά τα, την ε, τα κανάλια πληροφοριών. Εν μέρει συμφωνώ με τις τροπολογίες σας. Όμως δεν χρησιμοποιούν όλοι το διαδίκτυο. Πρέπει να συνεργαστούμε, να αντιμετωπίσουμε ε, τις ανισότητες ε, και να μην αποκλείσουμε αυτούς που δεν χρησιμοποιούν ε, την πληροφορική για πρόσβαση στις πληροφορίες. Έτσι λοιπόν πρέπει ο κλάδος να έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει έντυπο υλικό με δική του πρωτοβουλία και όχι μόνο κατόπιν ετήματος. Αυτό το σχέδιο πληροφοριών, το σχέδιο κειμένου πληροφοριών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από αίτημα του ε, κοινού ή μέσω των παρόχων ιατρικής ε, υγεία. Όσον αφορά τον έλεγχο των πληροφοριών, συμφωνώ ότι για πληροφορίε που δεν έχουν ακόμα εγκριθεί μέσω τη διαδικασία έγκριση αγορά, θα πρέπει να εγκρίνονται καταρχήν ω θέμα αρχή από τις αρμόδιε αρχέ. Όμω θα πρέπει να δώσουμε προσοχή και στα συνταγματικά ζητήματα που θέτουν κάποια κράτη-μέλη όσον αφορά τη ε, συμπατότητα με προκαταρ... του προκαταρτικού ελέγχου με την ελευθερία έκφραση. Θα πρέπει να υπάρχει εκ των υστέρων έλεγχο σχετικά με το ε, ε, ανάλογα βέβαια με το αν υπάρχει τέτοιου είδους έλεγχος. Όσον αφορά το αίτημα παροχής πληροφοριών από πηγές άλλες από ό,τι η βιομηχανία. Θέλω να υπογραμμίσω ότι συμφωνώ απόλυτα με την πολιτική φιλοδοξία οι προτάσεις να στηρίζονται σε, ε, στην βιομηχανία η οποία παρέχει τα φάρμακα όπως σήμερα και να υπάρχει μια ευρύτερη ε, ατζέντα για την ενημέρωση των ασθενών. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές πηγές που πρέπει να μελετηθούν ώστε δυνατόν καλύτερα καλύτερα. Οι παρούσες προτάσεις όμως δεν εμπίπτουν σε αυτό το τομέα. Πρέπει η Κομισιόν να ε, συντάξει προτάσεις για την αναγνωσιμότητα του ε, φυλαδίου του πακέτου. Είναι πρόωρο λοιπόν κάτι τέτοιο, ούτε θα ήταν σκόπιμο για κάθε κλινική μελέτη ε, που αναφέρεται στην, στην περίπτωση ε, στην περίληψη της ε, έκθεσης δεδομένων. Ένας ε, σύνδεσμος ηλεκτρονικά με τη βάση δεδομένων θα αρκεί. Όσον αφορά την, την έγκριση αγοράς και αυτή είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά. Όσον αφορά τώρα τις παροχές πληροφοριών από την βιομηχανία. Υπάρχουν κάποιες ιστοσελίδες και βάσει δεδομένων στην Ευρώπη που προσφέρουν τέτοιε πληροφορίες. Αυτό που δεν υπάρχει είναι η, η διασύνδεσή τους. Προτείνω να υπάρξει μια ε, ηλεκτρονική πύλη στην Ευρώπη ως ενιαία είσοδος για πρόσβαση αυτές τις πληροφορίες και γι' αυτό Αναγνωρίζω και την ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση για τι ασθένειε και τι διαστάσει του. Πρέπει οι ασθενεί να μάθουν όχι μόνο για τα φάρμακα αλλά και για τι εναλλακτικέ θεραπείες, εναλλακτικέ μορφές θεραπεία. Τέλο, η Κομισιόν βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να εξυπηρετήσει ένα ευρωπαϊκό τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωση. Ε, υπάρχουν και ε, τα κράτη-μέλη και οι οργανώσει ασθενών η, μπορεί να προσθεθεί αξία και πολλά ε, μέσα βοήθειας προς αυτήν την κατεύθυνση ήδη υφίστανται. Αγαπητά μέλη, δεν θα σας εκπλήξει ότι υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που, δεν μπορεί να υποστηρίξει η Κομισιόν μετά από σοβαρή μελέτη, ας πούμε, η, το δικαίωμα της... Ε, ε, ε, τη υποβολή παραπώνων υπάρχει ήδη και ισχύει και δεν χρειάζεται να αναδιατυπωθεί. Ένα κατάλογο τη θέση τη Κομισιόν επί όλων των ε, ε, τροπολογιών που προτείνονται έχει ήδη δοθεί στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα για μία ακόμα φορά να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και τον κύριο Φιέλνερ και του σκιώδη συζητητέ για την σημαντική του συνεισφορά. Ελπίζω ότι η ψηφοφορία αυτή την εβδομάδα θα ενισχύσει την πρόσβαση που θα έχουν οι ασθενεί πληροφορίε και θα πείσει το Συμβούλιο να ξεκινήσει μια σε βάθο συζήτηση των προτάσεων αυτών. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Επίτροπο. Επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Κορέιαντε Ντεκάμπο για την Επιτροπή ΙΤΡΕ. Ε, ε, Αγαπητέ Πρόεδρε, συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, ο ασθενή πρέπει να έχει δικαίωμα να ξέρει όσα περισσότερα γίνεται σχετικά με την ασθένειά του και με τα φάρμακα που υπάρχουν για την εντόπιση της όχι όμως διαφημιστικά. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε πώς λαμβάνει αντικειμενική ενημέρωση. Υπάρχει διαφορετική ερμηνεία των υφιστάμενων νομικών κειμένων, πρέπει να προσεγγιστούν μεταξύ τους και να ενισχυθεί η ενημέρωση του πολίτου. Η ενημέρωση πρέπει να είναι αξιόπιστη, προσπελάσιμη και να προσανατολίζεται προς ένα μέσο πολίτη που δεν είναι ειδικό να είναι αυτός ο πολίτης που τελικά αποφασίζει. Η προθεσμία που δόθηκε για την ε, σιωπηλή αποδοχή πρέπει να γίνει παντού 120 ημέρες. Η... Υπάρχει μία βασική πηγή ενημέρωσης που είναι οι ιατροί. Μια τελευταία η ιατροι μια τελευταια παρατηρηση Να συγχαρώ τον κύριο Φιέλνερ για τη δουλειά του και γιατί υιοθέτησε σχεδόν όλες τις προτάσεις τροπολογίες που υποβάλαμε ως Επιτροπή ε, Εσωτερικών, Εσωτερικής Αγοράς. Ο κ. Μπουσόη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Συγχαίρω και εγώ τον εισηγητή και τους συναδέλφους που συνέβαλαν στο φάκελο, στο θέμα αυτό και τον Επίτροπο κ. Ντάλη. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι καλό. Είναι πολύ πιο προσανατολισμένη προς τον πολίτη η έκθεση οι ασθενείς θέλουν όλο και περισσότερο να ενημερώνονται για να αποφασίζονται ενεργά στις αποφάσεις για την υγεία τους. Επίσης προσπαθούν να βρουν πληροφορίες online. Η ενημέρωση στο ίντερνετ δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Κάτι που δεν θα γίνει αν, δεν κάνουμε, αν μείνουμε αδρανείς. Πρέπει να μπορέσουμε να παρέχουμε νομοθεσία για την παρακολούθηση και έλεγχο των ε, ιστοσελίδων και την ε, πιστοποίηση κάποιων ιστοσελίδων για να ξέρει, για να είναι βέβαιος ασθενής για την πηγή της ενημέρωσης και για το κατά πόσον η ενημέρωση αυτή έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. Για τον σκοπό αυτό υιοθετήσαμε στην Επιτροπή μια σειρά ε, τροπολογιών ε, για την διαφήμιση, αλλάζοντας την λέξη διάδοση στο λέξη διάθεση, και ε, ε, ε, διευκολύνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης του ασθενού στην ενημέρωση όποτε και αν το χρειαστεί. Ευχαριστώ κύριε Μπουσόη. Οι αγορητές των πολιτικών ομάδων, ο κύριος Νέλχαρτ πρώτος για το ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, όταν σκεφτούμε ότι στην τελευταία θητεία συζητήσαμε αυτή την πρόταση της Επιτροπής και συζητήσαμε όλο το φάσμα από την πλήρη απόρριψη μέχρι την ε, επιβράβευση, θα πρέπει να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με αυτό το οποίο έχουμε τώρα ενώπιόν μας και γι' αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή γιατί από αυτό το μεγάλο φάσμα ε, απόψεων σε να παράγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η μαγική λέξη, η κεντρική λέξη είναι ο προσανατολισμός και η εστίαση στον ασθενή. Μας ενδιαφέρει αυτό το οποίο χρειάζεται ο ασθενής και πιστεύω ότι είναι σωστή η άποψη την οποία ακολουθούμε ότι μπορεί από ποικίλε οδούς, από ποικίλου διάβλους να πληροφορηθεί ο ασθενής και βέβαια θα παραμείνει ο γιατρός το άτομο εμπιστοσύνη του ασθενούς και βεβαίως θα επηρεάζει ο γιατρός τον ασθενή και αυτό το φροντίζουμε απαγορεύοντας τη διαφήμιση των φαρμακευτικών προϊόντων και οι πληροφορίες που φτάνουν στον ασθενή ελέγχονται και είναι εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές αξιολογούνται οι πληροφορίες επιστημονικά και είναι πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται ο ασθενής. Βεβαίω, οποιοδήποτε μπορεί να αναζητήσει πληροφορίε στο διαδίκτυο και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε γιατί αυτό το κάνουμε σε πολλού τομεί ε, και είναι κάτι το πολύ διαδεδομένο. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα έχει επιτέλου το θάρρο ε, να λάβει μέτρα για αυτή ε, την έκθεση. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δράσει γρήγορα γιατί είναι κάτι που το περιμένουν οι ασθενεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σνέλχαρτ. Ο κύριος Παγνιό εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτρόπε, αγαπητοί συνάδελφοι, στις αρχές του 21ου αιώνα οι ασθενείς έχουν τώρα ιδιαίτερα ανάγκη από τις κατάλληλες πληροφορίες για να μπορούν να συμμετέχουν οι ίδιοι την αγωγή τους και να αποφασίζουν μαζί με τους επαγγελματίες υγείας ποια θα είναι η αγωγή τους και για να, απο, να αποφασίσουν ότι θα ακολουθούν την αγωγή τους. Ζητούν οι ασθενείς πλέον ανεξάρτητες πληροφορίες που θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες όλων. Δυστυχώς η προτάση αναδιατύπωση της οδηγίας που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των πολιτών της Ευρώπης. Αυτές οι προτάσεις άνοιγαν το παράθυρο σε άμεση προώθηση προϊόντων από τις φαρμακευτικές εταιρείες, πράγμα το οποίο δεν ήταν καθόλου αυτό το οποίο θέλαμε για να ανταποκρινόμαστε στι ανάγκε των ασθενών. Αυτέ οι πληροφορίε δεν ε, είναι χρήσιμε ούτε για του πολίτε ούτε για τα κράτη-μέλη. Αντιθέτω, θα έδιναν περισσότερη, περισσότερη γραφειοκρατία, αύξηση των εξόδων και περισσότερου κινδύνου για του ασθενεί. Και γι' αυτό, καταρχήν, υποβάλαμε μια πρόταση απόρριψη ε, αυτού του κειμένου και ζητήσαμε από την Επιτροπή να επανεξετάσει την προσέγγιση τη και ήταν η θέση που υιοθέτησε ο Κάρλο Λούτερ, συνάδελφο από του Πρασίνου, και τελικά επέτρεψε στον κύριο Φιάλινα, στον εισηγητή, του οποίου χαιρετίζω την πρόταση, να περάσει σε μια συγκεκριμένη και πολύ σωστή εξέταση τη πρόταση τη Επιτροπή. Εξετάσαμε πολλέ τροπολογίε για να προστατεύσουμε το όφελο των καταναλωτών και για να διευκολύνουμε την πρόσβαση των ασθενών σε ανεξάρτητε και συγκριτικέ πληροφορίε που θα είναι προσαρμοσμένε στι ανάγκε του καθενό. Από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, η ε, ε, πρόταση τόνισε περισσότερο ε, την αναζήτηση των πληροφοριών από τους ασθενείς και όχι την προώθηση των πληροφοριών από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Αποφασίσαμε να αποσύρουμε την πρότασή μας για απόρριψη του κειμένου γιατί άλλαξε η ουσία του κειμένου προς τη σωστή κατεύθυνση τους τελευταίους μήνες. Το σχέδιο έκθεσης όπως έχει τροποποιηθεί κατορθώνει να αντισταθμίσει την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να αρνούμεθα το να ε, χειριζόμαστε τους επαγγελματίες υγείας ώστε ε, να προμηθεύουν στους στου ασθενείς τα φυλάδια που θα τους δίνουν οι φαρμακευτικές εταιρείε χωρίς κανένα έλεγχο από τις υπηρεσίες υγείας. Είναι σημαντικέ οι πληροφορίε, ιδίω σε τομεί όπω ο εμβολιασμός. Οι πληροφορίε δεν μπορούν να παρέχονται μαζικά από τις φαρμακευτικές εταιρείε. Πρέπει να, έχουμε, να είμαστε σε επαγρύπνηση Κλείνω κύριε Πρόεδρε και να μην ξεχνάμε αυτό που έγινε με το φάρμακο Μεντιδόρ που δείχνει πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε να υπάρχει σωστή ισορροπία, μια ισορροπία την οποία αναζητήσαμε με, αυτή την, το, με αυτό το σχέδιο έκθεση. Ευχαριστώ. Now, on of Liberal. Η κυρία Παρβάνοβα εκ μέρου των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ω ε, εκπρόσωπος του και ηγητή τη ομάδα μου θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Η, το κόμμα μας ε, θεωρεί ευπρόσδεκτη την έκθεση αυτή που ασχολείται με προβλήματα ε, των, της ενημέρωσης για τα φάρμακα. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια σαφής ε, σχέση πληροφοριών και των ασθενών και άρα θα πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος των πληροφοριών αυτών και αυτό θα πρέπει να υπάρχει μέσω στο σελίδων αλλά βεβαίως θα πρέπει να υπάρξουν και ασφαλιστικές δικλείδες για την παρακολούθηση και την ε, τήρηση της νομοθεσίας. Επίσης, Όσον αφορά το υλικό που προσφέρεται στους ε, επαγγελματίες της υγείας για την ενημέρωση, δεν υπάρχει ανάγκη να αποκλειστεί αυτό το υλικό από τις διατάξεις του υπόλοιπου περιεχομένου, γιατί εξ όσων γνωρίζουμε οι γιατροί είναι οι πιο έμπιστες πηγές, οι πιο αξιόπιστες πηγές πληροφοριών. Θα υποστηρίξω λοιπόν την τροπολογία 88 και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις βασικές βελτιώσεις που θα επιφέρει η έκθεση αυτή στην πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι υποστηρίζω την έκθεση. Καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μου ζωή υποστήριζα το δικαίωμα κάθε πολίτη να διαχειρίζεται την υγεία του. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σωστή ενημέρωση. Όπως είπε και ο κύριος Σνέλχαρτ, καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσης θητείας προσπαθούσαμε να προχωρήσουμε την ομοθεσία αυτή και, την, και να δια, η συζήτηση ότι δεν μπορεί να διακρίνουμε την ενημέρωση από την διαφήμιση είναι νόητη. Όλοι καταλαβαίνουμε τι είναι διαφήμιση και όλοι καταλαβαίνουμε τι είναι ενημέρωση. Ας καταλάβουμε λοιπόν ότι ζούμε σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Δεν μπορούμε να υποχρεώνουμε τους πολίτες της Ένωσης ε, να ψάχνουν πληροφορίες ε, σε αμερικανικές ε, ιστοσελίδες. Ας τους δώσουμε ευρωπαϊκές. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά. Ο κύριος Μασταλκα, 1,5 λεπτό. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως και ο συνάδελφος ο κ. Σούσκι, ήθελα και εγώ να πω ότι καθ' όλη την επαγγελματική μου σταδιοδρομία η προσπάθειά μου ήταν ε, προς την καλύτερη πληροφόρηση των ασθενών. Εκτιμώ ιδιαίτερα την προσπάθεια του εισηγητού να μια μικρή επιφύλαξη που θα εξηγήσω αργότερα. Όταν αρχίσαμε να συζητάμε το έγγραφο αυτό, είχαμε δύο προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Καταρχήν, δόθηκε ω αρμοδιότητα σε νέο επίτροπο και δεύτερον, έπρεπε να αποφασίσουμε αν θα συνεχίζαμε τη δουλειά μα πάνω στο προηγούμενο έγγραφο ή αν θα ξαναρχίζαμε από την αρχή. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ, ε, συμφωνήσαμε ότι η προηγούμενη πρόταση δεν ήταν σωστή, δεν ευθυγραμμιζόταν προ τα συμφέροντα των ασθενών και δεν θέλαμε να χάσουμε χρόνο. Ξεκινήσαμε λοιπόν να δουλεύουμε πάνω στο προηγούμενο έγγραφο. Συμφωνήσαμε ότι θα απορρίψουμε τις εμπορικές εκστρατείε. Ε, των φαρμακευτικών εταιριών. Θέλαμε να υπάρχουν έντυπα μέσα για τους ασθενείς και θα ήταν δικαίωμα των ασθενών να ζητούν πληροφορίες και θα έπρεπε οι ασθενείς να είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Μου κάνει εντύπωση που υποβάλλεται μια τροπολογία πάλι στην Ολομέλεια, η οποία απερίφθη στην Επιτροπή. Η έγκριση μια τέτοια τροπολογία θα ήταν ένα βήμα προ τα πίσω, πιστεύω. Αν εγκρίνουμε την πρόταση αυτή, εγώ θα έχω πρόβλημα στην υπερψήφιση του συνολικού κειμένου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την Ευρώπη, για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Ο κύριος Ρόσμπαχ, ένα λεπτό. Η κυρία Ρόσμπαχ, συγγνώμη. Πρόεδρε, συμφωνώ με τον εισηγητή. Η έμφαση πρέπει να είναι ασφάλεια και ενημέρωση για τον ασθενή. Οι επαγγελματίε της υγεία και οι ασθενεί πρέπει να έχουν την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στην ενημέρωση για κάποια φάρμακα. Κάποια φάρμακα μπορεί να θέλουν να έχουν, για κάποια φάρμακα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα ενημέρωσης των ειδικών. Χρειάζεται να υπάρχει λοιπόν ομοιόμορφη ε, περιγραφή των φαρμάκων, διότι συχνά ψάχνουν στο ίντερνετ για να βρουν ενημέρωση επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν τις ενδείξεις που περιλαμβάνουν οι οδηγίες του ή η δραστική ουσία του φαρμάκου. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε οι πληροφορίες αυτές να εξασφαλίσουμε ότι είναι ασφαλείς και να μην θεωρούνται ως μια μορφή διαφήμισης. Οι φαρμακευτικές εταιρείε, το ξέρουμε, πρέπει να πουλάνε τα προϊόντα τους. Ωστόσο η ευθύνη πρέπει να είναι εκεί που θα ενθαρρύνει την εμπιστοσύνη του πολίτη. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Για τους μη εγγεγραμμένους και για ένα λεπτό κύριο Σόμπερ Μάιερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στο επίκεντρο βρίσκεται το όφελος του καταναλωτού. Το καταναλωτή θέλουμε λοιπόν να προστατεύσουμε και οι φαρμακευτικές εταιρείες ε, τείνουν να παρέχουν στο φυλάδιο οδηγιών ε, πολύπλοκες πληροφορίες ε, που φοβίζουν τον καταναλωτή και δέχεται να αποτρέπουν τον καταναλωτή από τη σωστή λήψη των φαρμάκων του. Όσον αφορά την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, πρέπει να είναι τεκμηριωμένες οι πληροφορίες αυτές. Το φυλάδιο οδηγιών θα πρέπει να είναι ένα φυλάδιο προσαρμοσμένο στι ανάγκε του χρήστη, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο και ιδιαίτερα για του ηλικιωμένου ασθενείς θα πρέπει να παρέχει πληροφορίε ε, με τρόπο ε, εύληπτο. Ιδίως όσον αφορά και τις τρίτες χώρες, θα πρέπει να αποφύγουμε τις γκρίζες ζώνες και το παραεμπόριο. Ευχαριστώ. Ξεκινούμε την ε, συζήτηση με τους υπόλοιπους αγωγητές. Παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο σας, γιατί έχουμε καθυστερήσει και πρέπει να κλείσουμε πριν τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα δηλαδή. Ξεκινάμε με τον κύριο Ταταρέλα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η οδηγία που συζητούμε έχει στόχο να εναρμονίσει το περιεχόμενο και την ποιότητα των πληροφοριών φαρμακευτικού χαρακτήρα που είναι προσβατέ σε όλου του πολίτε τη Ένωση. Επαναλαμβάνοντα βεβαίω ε, την ε, αρχή τη διαφήμιση, καθιερώντα τόσο το δικαίωμα του ασθενού στην ενημέρωση. Πρέπει να δώσουμε σε όλου του Ευρωπαίου πολίτε την ίδια δυνατότητα πρόσβαση στην ενημέρωση για τα φάρμακα. Ο αρχικός στόχος της οδηγίας είναι να, να επιτρέψουμε στον πολίτη ασθενή να είναι περισσότερο ενημερωμένος και να μπορέσει έτσι να ε, αντιδράσει πιο ε, ε, συνειδητά στο φάρμακο. Όλοι και οι φαρμακευτικές εταιρείες ακόμα πρέπει να έχουμε τον ίδιο στόχο, τη διάδοση χρήσιμων και σωστών πληροφοριών ταυτόχρονα δε ε, χρήσιμων πληροφοριών για όλους τους πολίτες. Θεωρώ δύο τα σημαντικότερα σημεία της οδηγίας. Ένα, μέσω μιας σωστής ενημέρωσης δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα φάρμακα με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ούτως ώστε να βελτιώσει τα θετικά, τις θετικές συνέπειες στην υγεία, μειώνοντας ταυτόχρονα στο ελάχιστο τους κινδύνους από μια ε, λάθος χρήση τους. Δεύτερον, σωστή και αποτελεσματική ενημέρωση που μπορεί να αυξήσει στον πολίτη την επίγνωση του βάρους των φαρμακευτικών δαπανών στις γενικότερες δαπάνες. Ωστόσο, πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα. Ιδίως το κίνδυνο, η ενημέρωση για τα φάρμακα να γίνει και καλυμμένη διαφήμιση. Πρέπει να αποφύγουμε ε, να δίνονται κατ' επίφαση επιστημονικές πληροφορίες με στόχο να εξαπατηθεί ο ασθενής προς την, προς στόχο, με στόχο την αγορά ενός φαρμάκου. Υπάρχουν ευτυχώς ε, ικανοποιητικά μέσα ελέγχου, ιδίως αυτά που μπορεί να πάρει μέσω ίντερνετ ο ασθενής. Εύχομαι λοιπόν και κλείνω η Επιτροπή να προβλέψει τρόπους ενημέρωσης και ελέγχου των πληροφοριών τόσο ώστε να εξασφαλίσει την ορθότητά του Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να ανατεθούν σε οργανισμούς που, είναι, που έχουν αυτό το στόχο και είναι ανεξάρτητοι για να υπάρχει μεγαλύτερη αμεροληψία. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάντεμπαχ. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο Επίτροπος Ντάλι είπε ότι θα πρέπει να προσανατολιστούμε στον ασθενή και αν η πρόταση της Επιτροπής είχε στο επίκεντρο την αγορά, τώρα με πολλές τροπολογίες οι οποίες πέρασαν με μεγάλη πλειοψηφία, κατορθώσαμε να φέρουμε τον άνθρωπο στο προσκήνιο το δικαίωμα του ασθενούς ε, στις ε, αξιόπιστες πληροφορίες ε, που δεν θα διέπονται από την αρχή της προώθησης του προϊόντος αλλά από την αρχή της ζήτησης του, του προϊόντος είναι το σημαντικό. Προέρχομαι και εγώ από τον τομέα της διαφήμισης και ξέρω ότι η διαφήμιση έχει ως στόχο την πώληση. Εμείς όμως έχουμε το καθήκον να ενημερώσουμε και νομίζω ότι με την έκθεση που έχουμε ενώπιόν μας και με τις κατάλληλες τροπολογίες θα ανταποκριθούμε έχουμε σε αυτή την υποχρέωση που έχουμε, δηλαδή να παρέχουμε σωστή πληροφόρηση θέλουμε να είναι σωστά ενημερωμένοι οι ασθενείς και μέσω των φαρμάκων να, επιτύχουμε κατά προτίμηση την πρόληψη των ασθενειών και όχι την επιβάρηση των ασθενών με πολλά φάρμακα. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάννα Κουδάκη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πόσο συχνά αναρωτιόμαστε για τις ε, ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων που παίρνουμε, πόσο συχνά αναρωτιόμαστε ε, για τα διάφορα προϊόντα που δίνονται για τις διάφορες ασθένειες. Αυτά είναι προβλήματα που συχνά τίθενται και που δείχνουν το πόσο χρειάζεται το κοινό της πληροφορίας. Στην αρχική πρόταση του Συμβουλίου δεν υπήρχε η έμφαση στο δικαίωμα του ασθενούς για αναζήτηση πληροφοριών. αντιθέτω ήταν υποχρέωση των φαρμακευτικών εταιριών να παρέχουν πληροφορίε με απαγόρευση των διαφημίσεων για τα συνταχογραφούμενα φάρμακα επιτεύχθηκε αυτή η αλλαγή του στόχου και οι εθνικές αρχές και οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να είναι η βασική πηγή πληροφοριών και αυτό είναι κάτι το οποίο επετεύχθη. Η οδηγία για την πληροφόρηση των ασθενών δίνει ένα ισχυρό μήνυμα για τα δικαιώματα των ασθενών. Συγχαίρω τον εισηγητή διότι ασχολήθηκε με ένα δύσκολο θέμα και κατέληξε σε μια πρόταση συνεκτική που ελπίζω ότι όλοι θα υποστηρίξουμε ομόφωνα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάρκου Νάιτ, 1,5 λεπτό. Αγαπητέ κύριε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ συχνά υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών και των ασθενών και την ικανότητά τους να αναλάβουν μόνοι τους την υγεία, την υγεία τους. Εμείς όμως πρέπει ως πολιτικοί να προστατεύσουμε τους ασθενείς από ε, ανακριβείς πληροφορίες και γι' αυτό επιδιώκουμε μέσω αυτού του νομοθετήματος. Τώρα, η ενημέρωση για τα φάρμακα. Φαίνεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει μια μεγάλη ποικιλία καταστάσεων και δεν είναι ε, απόλυτα σαφές τι, ε, ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ τους. Γι' αυτό είμαι υπέρ του ξεκάθαρου καθορισμού των ενιών. Πρέπει για τον ασθενή να υπάρξουν αξιόπιστες ε, και αποτελεσματικές πληροφορίες ε, στη μητρική τους γλώσσα και προσβάσιμες από τους ασθενείς. Όσον αφορά τώρα το θέμα της κρυφής διαφήμισης, από αυτήν πρέπει να προστατεύσουμε όχι ε, τους ασθενείς, αλλά και τους πάντες και γι' αυτό επειδή όλοι οι εργονισμοί εξαφανίζονται πρέπει να διαφωτίσουμε περισσότερο την κατάσταση των ασθενών. Ελπίζω όλοι να είναι καλύτερα και σε καλύτερη υγεία. Ο κύριος Κάπερνοκ, ένα λεπτό. Πρόεδρε, η οδηγία για τα φαρμακευτικά προϊόντα είχε μείνει χωρίς αλλαγή για 10 χρόνια. Γι' αυτό ήρθε καιρό να την αλλάξουμε. Υποστηρίζω απόλυτα το δικαίωμα του ασθενή να ενημερώνεται πλήρω. Ταυτόχρονα πρέπει ο ασθενή να είναι πλήρω συμμέτοχος ε, στο, με το γιατρό στην λήψη των αποφάσεων. Να είναι και υπεύθυνο και να έχει γνώση. Βασικό ρόλο στην αλλαγή αυτή θα παίξει η διαθεσιμότητα της πληροφορίες που οι πληροφορίες όπως οι πληροφορίες για φαρμακευτικά προϊόντα και ακόμα και για τα φάρμακα που δίνονται μόνο με συνταγή. Ο ασθενής πρέπει να έχει πρόσβαση στην ε, ενημέρωση για τα φάρμακα και online και γραπτός που θα είναι αληθής, κατανοητή και ευανάγνωστη. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την δουλειά που έκανε. Έκανε πολύ καλή δουλειά και θα υποστηρίξω την πρότασή του. Και εμείς ευχαριστούμε. Η κυρία Βάις Γκέρμπερ. Ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον Κρίστοφερ Φιέλνερ και τον σκιώδη εισηγητή γιατί ήταν δύσκολες οι συνθήκες ε, και αντίξωες οι περιστάσεις και παρόλα αυτά κατέληξε σε πολύ καλό αποτέλεσμα την έκθεση αυτή. Η πρόταση της Επιτροπής βελτιώθηκε σημαντικά παραμένουμε στην απαγόρευση της διαφήμισης και δεν δίνεται πληροφόρηση ε, μέσω ε, ραδιοτηλεοπτικών μέσων και πρέπει οι ασθενείς να ζητήσουν τις πληροφορίες. Θέλουμε ασθενείς οι οποίοι να είναι υπεύθυνοι, ασθενείς οι οποίοι θα ζητούν τις πληροφορίες που τους χρειάζονται. Και γι' αυτό θέλουμε να μπαίνει ο ασθενής ε, στο προσκήνιο της πληροφόρησης. Θα ήθελα να τονίσω τα εξή σημεία. Και εγώ ασχολήθηκα στην ε, Επιτροπή Νέας Αγοράς, Εσωτερικής Αγοράς για ε, τη διαδικτυακή πύλη σχετικά με τα θέματα υγείας των καταναλωτών. Οι καταναλωτές πολύ συχνά βρίσκουν στο διαδίκτυο πληροφορίες που δεν είναι ε, ελεγμένες και εγκεκριμένες. Γι' αυτό θέλουμε να δώσουμε μια εναλλακτική λύση του να υπάρχουν εγκεκριμένες πληροφορίες. Ένα άλλο θέμα είναι η φαρμακοεπαγρύπνηση όπου υπάρχει και μια, μια διαδικτυακή σελίδα στην οποία υπάρχουν πληροφορίες που δίδονται στα διάφορα φάρμακα στο φυλάδιο οδηγιών. Θέλουμε να δίδονται σωστές πληροφορίες ε, για τις διάφορες ασθένειες για να επιτύχουμε και την πρόληψη των ασθενειών και αν σωστά κατάλαβα τον κύριο Επίτροπο ε, ε, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό αλλά θα ήθελα μια σαφή δήλωση του Επιτρόπου αν είναι ένα τομέα στον οποίο υποστηρίζετε και θα προωθήσετε. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκροστέτ. Ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Συγχαίρω τον εισηγητή μας κύριο Φιέρνα για την εξαιρετική δουλειά που έκανε εδώ και πολλούς μήνες για τις δύο αυτές εκθέσεις. Το λέω αυτό διότι χρόνια περιμέναμε τα κείμενα αυτά οι παλιότεροι εδώ θα θυμούνται ότι στην αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας θέλαμε να γίνει λόγος και για την ενημέρωση των ασθενών στα φάρμακα και τις θεραπείες, όμως δυστυχώς είχε υπάρξει σύγχυση μεταξύ διαφήμισης και ενημέρωσης. Σήμερα ωστόσο η ενημέρωση δεν πρέπει να επιτρέψει να υπάρχει και καλυμμένη διαφήμιση και στην έκθεση πλέον δεν υπάρχει δικαίωμα των επιχειρήσεων να ενημερώνουν, αλλά το δικαίωμα των ασθενών να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση. Άλλη λογική δηλαδή. Η προτεραιότητα είναι ο ασθενής και άλλωστε λέμε όχι στην ενημέρωση χωρίς αίτηση, κάτι που μειώνει τους διάβλους ενημέρωσης και άρα και τον κίνδυνο διαφήμισης. Οι ασθενείς θα πάνε οι ίδιοι να βρουν τις πληροφορίες που θέλουν, δεν τους επιβάλλουν οι διαφημίσεις στα περιοδικά, τις εφημερίδες, την τηλεόραση. Και αυτό διαφέρει από την διαφήμιση. Γι' αυτό χρειάζεται και ένας εκ των προτέρων έλεγχος κάποιων πληροφοριών που θα γίνεται από τις εθνικές αρχές Επίσης θα πρέπει να μπορούμε να επιτρέψουμε τη δημιουργία ε, site που θα είναι αντικειμενική αντικειμενικά και θα παρέχουν πληροφορίες και επί χάρτου και ηλεκτρονικά και όπου θα περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που θα είναι αντικειμενικές, σωστές, που περιμένουν οι ασθενείς εδώ και καιρό. Πρέπει το Συμβούλιο να αναλάβει τις ευθύνες του και να διαδεχθεί τη διαφήμιση αυτή. Δεν μπορούμε να έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση στις ιστοσελίδες. Δέκα χρόνια περιμένουμε να λάβει θέση το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κύρια Μεζάρος. Ενάμιση λεπτό. Ο κύριος Μεζάρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Φιέλνερ, γιατί χρειαζόμασταν μια τέτοια πρόταση για ένα κείμενο που θα δίνει καλύτερη πληροφόρηση στους ασθενείς, ιδιαίτερα για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ποιοτικέ οι πληροφορίες αυτές που θα δίνουν τη δυνατότητα στους ασθενείς να αντιμετωπίσουν ε, την ιατρική τους ε, κατάσταση και επίσης ο ασθενής θα πρέπει να είναι ενημερωμένος ε, και να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για την αγωγή του. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εδώ θέλουμε μέσω της σωστής ενημέρωσης του ασθενούς να παίξουμε και ένα σωστό ρόλο μέσω των φαρμακευτικών εταιριών που εδώ έχουν ένα σημαντικό ε, ρόλο. Συναντάμε πολλές δυσκολίες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της πληροφόρησης για τα θέματα των φαρμάκων. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπου δεν υπάρχει πρόσβαση ακόμη και σε στοιχειώδεις πληροφορίες και τελικά είναι πολλές οι ανισότητες στον τομέα της υγείας στα διάφορα κράτη-μέλη. Εκτός από την πληροφόρηση από το διαδίκτυο υπάρχουν και πιο παραδοσιακές μορφές πρόσβασης στην ενημέρωση, αλλά εδώ αποσκοπούμε όχι στο να ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις για τα δικαιώματά τους, αλλά ε, να ενημερώνουμε τους ασθενείς, να έχουν οι ασθενείς δικαίωμα στην πληροφόρηση και πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ πληροφόρησης και διαφήμισης. Και είναι σημαντική επίσης και η συνεισφορά των γιατρών, διότι ο θεράπων ιατρός είναι αυτός ο οποίος δίνει τη συνταγή και αυτός πρέπει να είναι η πρώτη πηγή πληροφοριών και γι' αυτό πρέπει να είναι η πρώτη και καλύτερη πηγή ενημέρωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα θα αρχίσουμε το Catch the Eye. Ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετίζω τη δουλειά του εισηγητή για την ποιότητα της ενημέρωσης των ε, φαρμάκων ε, για τα φάρμακα των ασθενών. Ως γιατρός αντιλαμβάνομαι ότι η ενημέρωση για τα φάρμακα είναι εύληπτη από τους γιατρούς αλλά πρέπει να συμβεί το ίδιο και με τους ασθενείς. Υπάρχει και η διαδικτυακή διαφήμιση η οποία είναι παραπλανητική ή εσφαλμένη και μιλάμε για φάρμακα που διαφημίζονται μέσω διαδικτύου και τα οποία όχι απλώς δεν θεραπεύουν, αλλά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη. Για μία ακόμα φορά θέλω να υπογραμμίσω ότι η απάντηση εδώ είναι να εφαρμοστεί όλο το δυνατόν ε, γρηγορότερα η καλή πρόταση, η πρόταση που έχουμε υποβάλει για το ε, ε, σήμα αξιοπιστία. Και μόνο έτσι θα μπορέσει να υπάρχει αξιόπιστο και ασφαλέ περιεχόμενο και ήδη αυτό υπήρχε στο, στην έκθεσή μου για τους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Πυρίλο, ένα λεπτό. Πρόεδρε Επίτροπε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, η έκθεση που συζητούμε, οι εκθέσει που συζητούμε είναι πολύ σημαντικέ, διότι επιτρέπουν την εναρμόνιση τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την πρόσβαση στι πληροφορίε για τα φάρμακα, ιδίω διότι θα εξασφαλίζει το δικαίωμα ενημέρωση των ασθενών για τα φάρμακα και τα συνταγογραφημένα. Οι πληροφορίες αυτές ε, πρέπει να είναι ανεξάρτητες και να παρέχουν διαφάνεια για να εξασφαλίσουν ότι ε, παρέχονται και ελέγχονται όλες οι πληροφορίες από τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές απο, αποφεύγοντας έτσι να γίνουν ε, και καλυμμένη πρόθεση των φαρμάκων προς όφελος των επιχειρήσεων. Ζητώ επίσης την ίδια προσοχή και για τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται τα, οι οδηγίες των συνταγογραφημένων ε, ε, φαρμάκων. Σε μια τέτοια περίπτωση καλύτερα θα είναι για το, οι γιατροί ή οι φαρμακοποιοί που θα ενημερώνουν λεπτομεριακά τον ε, ασθενή για να υπάρχει πλήρης επίγνωση για το περιεχόμενο των φαρμάκων που παρέχονται. Ο κύριος Ρώση, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ο κανονισμός είναι θετικός. Ο στόχος του είναι να παράσχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που είναι εναρμονισμένο για τις πληροφορίες μη διαφημιστικού χαρακτήρα για φάρμακα που υπάρχουν στη συνταγράφηση, που μπορούν να παρέχουν στο κοινό οι φαρμακευτικές εταιρείες διαφυλάσσονται ωστόσο την απαγόρευση διαφήμιση. Αυτή η διαφοροποίηση διαφήμισης και ενημέρωσης είναι σημαντική. Βασίζεται στην αρχή της ενεργού έρευνας. Η έρευνα, η ενημέρωση για τα φάρμακα πρέπει να παρέχεται κατά βάση από τους γιατρούς. Οι υπόλοιπε πληροφορίες είναι συμπληρωματικές, πρέπει να, να διατηρήσονται, αλλά πρέπει να αποφεύγονται οι, οι ιατρικές ε, επιθεωρήσεις. Η ενημέρωση του ασθενούς με την ενεργή συμμετοχή του και των ε, επιχειρήσεων, ε, των οργανώσεων πολιτών είναι σημαντική και η ψήφος είναι υπέρ. Η κυρία Μαγκίνε, τελευταία ομιλήτρια για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όλοι επιθυμούμε οι ασθενείς να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτούς. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι τη χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών. Συμφωνώ ε, με τους συναδέλφους που λένε ότι δεν πρέπει να διαφημίζονται τα προϊόντα, αλλά επίσης πρέπει να πω ότι η μετάδοση υψηλή ποιότητα ε, πληροφοριών στους ασθενείς είναι η καλύτερη διαφήμιση, γιατί αυτό είναι ξεκάθαρο ε, μήνυμα που πρέπει να στέλνετε όπου χρειάζεται πρέπει λοιπόν οι γιατροί να να μεταδίδουν επιστημονικές πληροφορίες στους ασθενείς τους. Αυτό πολύ συχνά δεν γίνεται. Επίσης, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το, τον τρόπο με τον οποίο τα φάρμακα θα κατανέμονται, σε, αν θέλετε να το πω έτσι, σε ασθενείς διαφόρων ηλικιών. Σήμερα ε, είναι ένα θέμα που δεν έχει εξεταστεί για πάρα πολλά χρόνια. Είναι, πρέπει να δούμε με πολύ περισσότερο εμπιστατωμένο τρόπο πώς παρέχεται η περίφερψη στους ασθενείς. Ο Επίτροπος κ. έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι με ικανοποιεί που βλέπω τόσο μεγάλο βαθμό θετικής, ε, ε, θετικού ενδιαφέροντος για ένα νομοθέτημα και μια γενική συμφωνία που αφορά την ε, εμπιστοσύνη που υπάρχει για τις βασικές αρχές και τις έννοιες που περιλαμβάνει αυτή η πρόταση, όπως είπα και προηγουμένως. Ήταν πολύ σημαντικό να μεταφερθεί το επίκεντρο της αρχικής πρότασης προς τους ασθενείς. Να γίνει μια πρόταση που να στηρίζεται, στο, που να επικεντρώνεται στους ασθενείς. Έχω παρακολουθήσει ε, πολύ προσεκτικά τη συζήτηση που πραγματοποιείται στο Κοινοβούλιο. Έχω έρθει και σε επαφή με κάποιους από εσά για να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις και οι σκέψεις σας. Και όπως είπα και στην αρχική μου ομιλία, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά θετικό, επί του οποίου πρέπει να οικοδομήσουμε εν ώψη μιας τελικής συμφωνίας. Θα ήθελα να σχολιάσω εν συντομία αυτά που είπατε κι εσείς. Δηλαδή, εκ των ε, προτέρων έλεγχος που ανέφερε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό είναι λίγο υπερβολικές οι 120 μέρες κατά τη γνώμη μου. Εμείς θα προτείνουμε μάλλον κάτι γύρω στις 60 μέρες. Το διαδίκτυο, τεράστιο έργο. Ο έλεγχος των ιστοσελίδων που, που στέλνουν πληροφορίες στους ασθενείς είναι ζωτική σημασία. Όλοι όμως αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και δύσκολο. Τα θέματα που έθεσαν ο κύριος Μπουζό και η κυρία Γκροστέτ για τους ε, κανόνες, τους αυστηρούς κανόνες που θα διέπουν το διαδίκτυο είναι πολύ σημαντικό και προς τα εκεί πρέπει να κινηθούμε. Επίσης, το επίκεντρο, ότι δηλαδή ο γιατρός πρέπει να συνεχίσει να έχει ε, επικοινωνία με τον ασθενή, όπως ε, ανέφερε ο κύριος Σνέλχαρτ, πολύ σημαντικό. Και όπως επίσης το ανέφεραν ο κύριος Περνό και η Παρμάνοφ. Βεβαίως δεν θα πρέπει οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τους γιατρούς. Από την άλλη όμως πλευρά πρέπει οι γιατροί να αποτελέσουν ένα σωστό μέσον ροής των πληροφοριών. Εδώ πρέπει να εξασφαλίσουμε για μία ακόμα φορά ότι οι πληροφορίες που φτάνουν στα χέρια των γιατρών, όπως είπε και η κυρία Ρόσμπακ, θα πρέπει να είναι και αυτές αντικειμενικές. Τελευταίο σημείο σχετικά με την ολοκληρωμένη διαδικτυακή πύλη για τις ασθένειες που ανάφερε η κυρία Βουεσκρέμπερ. Πρέπει να πω ότι όσον αφορά τα φάρμακα, ήδη προβλέπεται κάτι τέτοιο από την ομοθεσία της φαρμακοεπαγρύπνησης την οποία προτείνουμε. Για τις ασθένειες τα πράγματα όμως είναι λίγο πιο δύσκολα. Ήδη Υπάρχει μια διαδικτυακή πύλη για τις σπάνιες παθήσεις. Όμως γενικά για το σύνολο των ασθενειών έχουμε ξεκινήσει και επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα, το οποίο όμως αποδεικνύεται εξαιρετικά σύνθετο και όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια εξαιρετικά εκτεταμένη ε, επιχείρηση. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους για τη δουλειά που κάνατε ε, στο θέμα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή, τους συνεισηγητές ε, για το έργο τους και όπως σας είπα ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα έγγραφο επί το οποίο θα μπορούμε να δουλέψουμε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Ο εισηγητής κ. Φιέλνερ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που ξεκίνησε η Κομισιόν ε, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσβαση στις πληροφορίες για τα φάρμακα διαφέρει πολύ ανά την Ευρώπη. Πράγματι, είναι καλό να έχουν όλοι πληροφορίες για τα φάρμακα. Και εγώ είχα και εγώ κάποιες απαιτήσει, δηλαδή να μην υπάρχει χώρα που η κατάσταση να επιδεινωθεί οι κάτοικοι της Σουηδίας ανησυχούν από αυτού γιατί επί χρόνια υπάρχει ένα σύστημα στη Σουηδία και πρέπει να πω ότι θα επιτραπεί το σύστημα αυτό, το φάσο όπως ονομάζεται, να διατηρηθεί στη Σουηδία και άλλες χώρες να εισάγουν ε, άλλα συστήματα, ε, παρόμοια συστήματα. Αν δείτε την κατάσταση σήμερα στην Ευρώπη, οποιοδήποτε θέλει να πει οτιδήποτε για ένα φάρμακο μπορεί να το κάνει πέρα από τις εταιρείε οι οποίες και αυτές, αυτές κατασκευάζουν τα, προβλήματα, τα, τα φάρμακα και οι οποίες ξέρουν τα περισσότερα εννοείται. Χαίρομαι λοιπόν που σήμερα ξεκινήσαμε την ιδέα της υποχρέωσης που θα έχουν οι φαρμακευτικές εταιρείες να δημοσιεύουν πληροφορίες για τα φάρμακα που παράγουν. Χαίρομαι επίσης που για όλα τα βασικά σημεία της ε, έκθεσης συμφωνείτε και εσείς και εγώ κύριε Επίτροπε. Υπάρχει ε, ενότητα Κοινοβουλίου και Κομισιόν και άρα θα ασκηθεί σοβαρή πίεση επί του Συμβουλίου για σοβαρή δουλειά. Ε, νομίζω ότι και στα σημεία επί των οποίων έχει φυλάξει η Κομισιόν, εμείς ε, είμαστε πολύ κοντά σχετικά με το έντυπο υλικό, ας πούμε. Υπάρχουν χώρες τις οποίες υπάρχουν ε, συνταγματικά προβλήματα επ' αυτού, όπως η Σουηδία. Παρά τα αυτά όμως πιστεύω ότι η θέση μας είναι πολύ κοντά. Υπήρξαν συνάδελφοι που είπαν ότι πρέπει να υπάρξει εξαίρεση για τις πληροφορίες που παρέχουν οι γιατροί. Θεωρώ ότι ένας γιατρός που βλέπει μια κλινική μελέτη δημοσιευμένη από μια εταιρεία θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να τη δώσει σε έναν ασθενή που θεωρεί ότι τον αφορά. Ή επίσης ένας ασθενής που βρίσκει το φυλάδιο ενημέρωση των ασθενών σε άλλη γλώσσα έχει το δικαίωμα να το δώσει στον ασθενή του. Πρέπει λοιπόν πράγματι οι γιατροί να μπορεί να αποφασίσουν τι δίνουν ω ενημερωτικό υλικό στου ασθενεί. Είναι πάντοτε ευθύνη των γιατρών και εδώ εμεί δεν πρέπει να παρέμβουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώθηκε εκείνη η συζήτηση. Η πληροφορία θα γίνει την Τετάρτη στις 12.